Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη για τη μικρή διακοπή, αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που είμαστε έτοιμοι για την ώρα των ερωτήσεων, τσακ στην ώρα της. Ακριβώς το επόμενο θέμα είναι πράγματι οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Και η πρώτη ερώτηση <clears throat> είναι από τον κύριο Μπέρντ Πόσελ και αφορά αυτό τις εθνοτικές μειονότητες στη Σερβία. Έχετε το λόγο κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Πόσελτ για το ερώτημα το οποίο έθεσε. Οι συνεδρία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 7 και 8 Δεκεμβρίου εφέτος ενέκρινε μία σειρά συμπερασμάτων για την ε, διεύνηση και τη Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και Σταθεροποίησης με τα Βαλκάνια. Το Συμβούλιο καλωσόρισε την δέσμευση της Σερβίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το έργο το οποίο λαμβάνει η χώρα για να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις και προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και τόνισε το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να τηρηθεί η ημερήσια διάταξη για την μεταρρύθμιση. Στις 14 Οκτωβρίου επίσης είχαμε μια ανακοίνωση τύπου η οποία περιέγραφε το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της δικαιοσύνης στην Σερβία και το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τύχουν απόλυτης απόλυτου σεβασμού στην Σερβία. Ο νέο Υπουργό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι μειονότητε στη Σερβία θα διδραματίσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτά. Χρειάζονται όμω να γίνουν περισσότερα για να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για την ανάγκη εφαρμογή των διεθνών προτύπων στη Σερβία και το Συμβούλιο τόνισε το γεγονό ότι η Σερβία έχει κυρώσει τα πιο σημαντικά ε, διεθνή μέσα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σερβία. Σε ό,τι αφορά την Νότια Σερβία και την κατάσταση που επικρατεί εκεί, όπω υπέδειξε το αξιότιμο και έντιμο κύριο μέλο, είναι γεγονό ότι υπήρξαν γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα τον Ιούλιο και συνελήφθησαν ορισμένοι από του δράστε. Μετά όμω από αυτέ τι συλλήψει, η κατάσταση, από ό,τι φαίνεται στη Νότια Σερβία, έχει βελτιωθεί. Οι πιο σημαντικές εθνικές ομάδες της αλβανικής ιδίως κοινότητας συμμετέχουν στο έργο του Συμβουλίου Συντονισμού και στις προσπάθειες για την διεύρυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ανοίξει ένα ειδικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Μετόκια που διδάσκει και σερβικά αλλά και αλβανικά και θα υπάρξουν περαιτέρω ε, θεσμοί και ενώσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν για να προωθήσουν τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα. Είναι ακόμα ασθενεί οι δομέ στην περιοχή αυτή και αυτό δημιουργεί προβλήματα για τι εθνοτικέ ομάδε στην Νότια Σερβία, η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδίω θα δώσουν μεγάλη σημασία στην κατάσταση αυτή τη Σερβία και θα προσπαθήσουν να προωθήσουν την ειρήνη και σταθεροποίηση τη περιοχή σε στενή συνεργασία με τη σερβική κυβέρνηση και του τοπικού πολιτικού ηγέτε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πόσσελτ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο καλή σας απάντηση. Αλλά έρχεται τις περιοχές αυτές τις συ... συνοριακές στην Σερβία, στην νότια περιοχή, τη Βοηβοδίνα και το Πρέσεβο. Θα πρέπει εσείς ως Επίτροπος λοιπόν να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι περιοχές θα τύχουν ανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων διαμεθοριακού χαρακτήρα και μέσα στη Σερβία, στο Σαντζάκι του Νόβι Παζάρ, υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά των μειονοτήτων πρέπει να εξασφαλιστεί και η οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει ακόμα μεγάλη βία στην Σερβία και ζητώ από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει αυτή την δυνητικά εκρηκτική κατάσταση. Υπουργέ. Κύριε Πόσελτ, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης ε, ούτως ή άλλως ε, και η Κομισιόν θα κάνει το ίδιο. Ε, η κατάσταση είναι ακόμα λεπτή, αλλά σίγουρα υπάρχει βελτίωση της κατάστασης και αυτό είναι αισιόδοξο για το μέλλον. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή, προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Όβερμαϊερ θέλει να παρέμβει για αυτό το θέμα. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει και στο Κωσυφοπαίδιο βία και όχι μονάχα στη Σερβία. Από τη μια μεριά έχουμε την αλβανική μειονότητα στη Σερβία, από την άλλη μεριά έχουμε τη σερβική μειονότητα στο Κωσυφοπαίδιο. Πού βρίσκεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν φαιές ζώνες και ασάφεια. Όταν έχουμε καταπιέσεις εθνοτικών ομάδων, θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από τη δική μας πλευρά και όλα αυτά δεν πρέπει να αναμειχθούν με το θέμα της αναγνώρισης του Κωσυφοπέδιου ως ανεξαρτήτου κράτους. Η κυρία Υπουργό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν κατανόησα ακριβώ πού ευρίσκεται το ερώτημα. Για το Κωσυφοπέδιο φυσικά γίνονται ε, εργασίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το γεγονό ότι δεν έχουν αναγνωρίσει όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Κωσυφοπέδιο, αλλά γίνονται προσπάθειε από την πλευρά τη Κομισιόν για να δούμε πώ μπορούμε να διευκολύνουμε την αντιμετώπιση των αθλητικών θεμάτων και στο Κωσυφοπέδιο. Παραμένουν δυσκολίε επιτοπίω, αλλά θα υπάρξει και στο μέλλον η διευκόλυνση για τι προξενικέ θεωρήσει. Αν αυτό εννοούσε ο αξιότιμο κ. Βουλευτή. Νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε λιγάκι από το κύριο θέμα, αλλά συνδέεται και αυτό με αυτό. Ε, το επόμενο ερώτημα το έχει υποβάλει η κυρία Χάρκιν και αφορά την ανεργία και τα επίπεδα ανεργίας. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο, όταν είστε έτοιμοι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν, για το ερώτημα αυτό. Η σημερινή κρίση φυσικά είχε επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους και τους έπληξε πολύ άσχημα. Ε, είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις οικονομική κρίσης. Θα πρέπει να σκεφτούμε τη γύρανση του πληθυσμού. Ε, τα κράτη-μέλη ακριβώς θα πρέπει να μειώσουν τα επίπεδα ενεργείας τους και να προσπαθήσουν να, να προσπαθήσουν να αποφύγουν τη διαιώνιση τη ανεργία. Φυσικά τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την πολιτική του απασχόληση, αλλά το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόληση ε, έχει υιοθετήσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ πριν από λίγα χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι δεδομένων των διαφορών στην αγορά εργασία στα διάφορα κράτη-μέλη και τα μέτρα θα πρέπει να είναι προφανώ διαφορετικά. Ε, έχουμε συντάξει μια κοινή έκθεση για αυτό το θέμα και το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, μιλάνε για την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Με τη σημερινή κατάσταση ε, έχουμε τονίσει ε, ποια είναι η κατάσταση της ανεργίας. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανάκαμψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τονίσαμε αυτό το Δεκέμβριο. Ε, και έχουμε δημιουργήσει και ένα πλαίσιο για τα μέτρα που θα υιοθετηθούν. Τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν ένα, ψήφισμα για τις αλλαγές που θα πρέπει να προωθήσουμε για να καταπολεμήσουμε την κρίση. Υπάρχουν διάφορες, διάφορα μέτρα ανάλογα με την εκάστοτε εθνική κατάσταση. Ε, θα μπορούσαμε ας πούμε να προσαρμόσουμε το χρόνο εργασίας τόσο ώστε να μειωθούν οι συσφορές. Ε, θα μπορούσαμε να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Θα μπορούσαν οι αρχές ε, να βελτιώσουν την κατάσταση της εργασίας των νέων Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση του ε, Συμβουλίου. Μετά, μετά την Σύνοδο Κορυφή του Ιουνίου, το Συμβούλιο επίση μίλησε για διάφορα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη και του εταίρου στην αγορά εργασία για να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει τη κρίση. Με την εισαγωγή τη αρχή τη ασφαλη ευελιξία, flexicurity ευέλικτος χρόνο εργασία, Αυτό νομίζω βελτιώνει την κατάσταση για τους επιχειρηματίε και ελπίζω τελικά θα οδηγήσει σε μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε περισσότερα κίνητρα, να μειώσουμε το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη των εισοδημάτων και διευκόλυνση της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας. Οι Υπουργοί γενικά συμφώνησαν ότι μια ενεργός πολιτική επασχόλησης με βραχυπρόθεσμα μέτρα θα πρέπει να προωθηθούν ε, κατάρτιση, εκπαίδευση, τέτοια μέτρα τα οποία ε, ξαναβάζουν τον κόσμο μέσα στην αγορά εργασία. Επίση, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η απασχόληση είναι πολύ σημαντικό παράγοντα για να αποφευθεί ο αποκλεισμό. Ε, υπάρχει σχέση μεταξύ τη απασχόληση, τη ε, ισότητα Γι' αυτό τα κράτη-μέλη ε, ενθαρρύνονται για να βελτιώσουν ε, και όλο το σύστημα των παιδικών σταθμών, ε, τη μείωση των ασυνσοτήτων στους μισθούς γυναικών και ανδρών. Υπάρχουν πάρα πολλά ειδικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά. Την απασχόληση των ηλικιωμένων, τα άτομα ανάγκες και τους νέους φυσικά. για την περίοδο 2010-2018. Αυτό το αρχικό πρόγραμμα υιοθετήθηκε από την Κομισιόν το 2009. Ευχαριστώ, η κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ ε, για την απάντησή σας, κυρία Μάλστρομ. Χαίρομαι που σας βλέπω και ελπίζω να σας ε, βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια και να απαντάτε σε ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Δύο σχόλια νομίζω πρέπει να κάνω. Δεν τα αναφέρατε στην απάντησή σας. Καταρχά θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα. Και δεύτερον, να αυξήσουμε ε, την, ε, τις δαπάνες στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Μέχρι στιγμή ε, είχαμε βασιστεί την ανοιχτή μέθοδο του συντονισμού. Είναι ένα ασθενικό μέσο και εργαλείο. Νομίζω ότι δεν τα καταφέραμε για να πετύχουμε τους στόχους της ατζέντα της Λισαβόνας. Ε, πώς θα ενδυναμώσετε αυτό το μηχανισμό, έχετε κάποιες ιδέες. Υπουργός ενδιαφέρουσα ερώτηση. Το Συμβούλιο μετά την πρόταση της Κομισιόν άρχισε να συζητάει το μέλλον της στρατηγικής της Λισαβόνας, ε, η Ευρώπη του 2020. Αυτό θα αποφασιστεί αργότερα επί Ισπανικής Προεδρίας, την Άνοιξη κάπου. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα βγούμε από τη σημερινή κρίση μακροπρόθεσμα, πώς θα δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, πιο επιχειρηματική Ευρώπη, πώς θα αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία, πώς θα επενδύσουμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη, ούτως ώστε η Ευρώπη να είναι πραγματικά δυνατός παγκόσμιος εταίρος στη διεθνή οικονομία. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στη νέα στρατηγική. Και ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής είναι η μέθοδος που επιλέγουμε. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί, θα πρέπει να εμπλέξουμε περισσότερο τι τοπικέ και περιφερειακές αρχές, γιατί αυτοί ουσιαστικά εφαρμόζουν τη μέθοδο. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και η εθνική ιδιοκτησία των προγραμμάτων, γι' αυτό εξετάζουμε και τον governance. Όλα αυτά τα εξετάζουμε και τα λέμε στο κείμενο τη Κομισιόν ε, και τώρα είμαστε στη φάση των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω θα προκύψουν καλέ προτάσει, γιατί πραγματικά έχετε δίκιο ότι είναι ένα από τα αδύναμα σημεία τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Ο κ. Μάτσα και ο κ. Ρουμπίκ θα μιλήσουν για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, κύρια Πρόεδρε. Αναφέρθηκε το λεγόμενο εργαλείο της μικροχρηματοδότησης και θα έρθουν τα χρήματα γι' αυτό από το πρόγραμμα Progress. Πώς θα εξασφαλιστεί όμως ότι αυτό το νέο μέτρο δεν θα λειτουργήσει σε βάρος ήδη αποφασισμένων προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής υποστήριξης. Ευχαριστώ κύριο Ρούμπικ. Κυρία Πρόεδρε, το ερώτημά μου ακολουθεί την εξή ε, κατεύθυνση. Μήπως είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ανέλθει και η ανεργία. Και αυτό βασίζεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι νεοστοί, δημιουργηθήσεις. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν βάσει των βελτίστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς οι οποίοι δημιουργούν νέες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας είπα ότι η τελική ευθύνη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι των κρατών μελών φυσικά. Αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά και όπως είπα στην αρχή προς την κυρία Χάρκινγκ έχουν υπάρξει συστάσεις του Συμβουλίου για το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ευελιξία ως προς την απασχόληση, τα διάφορα συστήματα στήριξης ώστε να αποφευθούν οι μηχανισμοί του αποκλεισμού και πρέπει να συνεχιστούν τέτοιου είδους συνεννοήσεις σε υψηλό επίπεδο με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κυβερνήσεις για να υπάρξει και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Πρέπει να δώσουμε ο ημέν στους δε παραδείγματα για να βρεθούν οι καλύτεροι τρόποι επίλυσης. Υπάρχουν οι συστάσεις λοιπόν του Συμβουλίου αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ε, πληρέστερα, ανάλογα με τις συνθήκε που ισχύουν στην καθεμία βέβαια, στο καθένα. Κατά τα άλλα δεν είμαι σίγουροι ότι κατάλαβα καλά την τελευταία ερώτηση, ίσως υπήρξε μεταφραστικό πρόβλημα, εγώ δεν μίλησα για μικροευθύνες, μίλησα για γενικό συντονισμό, για περισσότερη ευελιξία για περισσότερη συνεννόηση εταιριών και κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίε με τους απολυωμένους ή τους ανέργους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Επόμενο ερώτημα του κυρίου Σβάντσης ή Χουντή. Χουντή, Χουντή. Τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία το θέμα της μετανάστευσης είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εταιρικές σχέσεις με τις ε, με τρίτες χώρες ως προς τους ελέγχους στα σύνορα και για να υπάρξει ολοκληρωμένος έλεγχος στα σύνορα που ενέκρινε το Δεκέμβριο 2006 το Συμβούλιο θα ήθελα να πω ότι εφαρμόζεται συνεργασία με τις χώρες προέλευσης μεταναστών και είναι σημαντικό τμήμα αυτό των εργασιών του Frontex το οποίο έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει συνεργασία με τρίτες χώρες στα πλαίσια της πολιτικής της Ένωσης για τη μετανάστευση γενικότερα και στα πλαίσια όμως επίσης διμερών συμφωνιών. Ήδη έχουν γίνει, οργανωθεί τέτοιες συνεννοήσεις και συνεννοήσεις και η εντολή που ισχύει περιλαμβάνει και συναντήσεις με τουρκικές αρχές. Επειδή όμως δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι διαπραγματεύσεις αυτές, δεν μπορεί το Συμβούλιο να σας σχολιάσει πληρέστερα τι θα γίνει τελικά. Ευχαριστούμε ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, από τη σημερινή σας απάντηση καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τρία σημεία. Το πρώτο ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Frontex και της Τουρκίας βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο το δεύτερο ότι οι διαπραγματεύσεις είναι σε γνώση φαντάζομαι όλων των μελών της ευρωπαϊκής ένωσης και επομένως και της ελλάδας και επίσης ότι από τα συμπεράσματα της πρόσφατης συνόδου των υπουργών εξωτερικών η συμφωνία επανεισδοχής συνδέεται με τον έλεγχο των συνόρων. Αν είναι έτσι τα πράγματα, η Τουρκία δηλαδή ζήτησε για να συνεργαστεί για τη συμφωνία επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή επιχειρησιακή έρευνα με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε πώ ξεπερνιέται το σοβαρό θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των μεταναστών και το ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα όχι τόσο του ελέγχου των συνόρων όσο του ορισμού των συνόρων. δέχεται δηλαδή η τουρκία τα εξωτερικά σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης; δέχεται ότι η frontex ενεργεί επί των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς αυτό είναι ένα αχανές θέμα και οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έχουν μόλις ξεκινήσει. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος ε, Μπαρό και ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Μπίλστρομ, είχαν δείξει το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν ξεκινήσει προφανώς οι συζητήσεις, αλλά δεν έχουν αποδώσει ακόμα καρπούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας κρατούμε ενήμερους γιατί συνεχίζονται αυτές οι συζητήσεις και όλα τα κρατημέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα θα είναι πλήρως ενήμεροι για αυτές τις συζητήσεις. Και είναι απαραίτητο να τονιστεί ο σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες σε αυτές τις συνομιλίες, επομένως δεν χρειάζεται να ελέγξετε ότι αυτό θα συμβεί, είναι προφανές. Αλλά οι συζητήσεις αυτέ έχουν ξεκινήσει, προχωρούν, δεν έχουν περατωθεί, αλλά συζητούμε ακόμα. Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετέχουν και φυσικά εφόσον και η Ελλάδα συμμετέχει στη Frontex είναι και αυτή μέσα σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Δύο αιτήσει για συμπληρωματικά ερωτήματα. Σας πενθυμίζω δύο μονάχα πράγματα. Πρώτον, ότι οι συμπληρωματικές ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται σε 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι τώρα έχουμε πάει πολύ καλά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. <clears throat> Και δεύτερον, μόνο δύο συμπληρωματικές ερωτήσει σε μία ώρα των ερωτήσεων μπορείτε να θέσετε. Ο κ. Παπα-Νικολάου λοιπόν και ο κ. Λότσε. Κ. Παπα-Νικολάου πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η, συνεννο... συνεννόηση που κάνουμε με την Τουρκία για την τελική κατάληξη σε συμφωνία επανεισδοχής για τα θέματα της μετανάστευσης θα περιλαμβάνει και ζητήματα σε σχέση με τη συνεργασία για τη frontex. και το δεύτερο που θέλω να πω εμείς έχουμε διαπιστώσει στην ελλάδα το τελευταίο διάστημα παρενοχλήσεις των αεροσκαφών της frontex από τις τουρκικές αρχές. Ε, στις απαντήσεις της κομισιόν δεν έχουμε πάρει συγκεκριμένη ε, απάντηση σε ό,τι αφορά ε, την επικοινωνία που γίνεται και αν αυτό τελικά συνιστά παρενόχληση. αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού. ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ χωρίς μικρόφων. Σίγουρα είναι σημαντικό να υπάρξει διεθνή συνεργασία, αλλά δεν έχει νόημα αυτό όταν αυτή η συνεργασία τρίτων χωρών πρέπει να εξαγοριστεί με την οικονομική βοήθεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες συνεργασίες οι οποίες προβλέπονται και δίνεται πράγματι κάποιο οικονομικό κίνητρο στην Τουρκία να συνεργαστεί με τη Frontex ή όχι. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα των ε, σκαφών της Frontex έχει τεθεί πολλές φορές στην ώρα ερωτήσεων και οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν τονίσει στις τουρκικές αρχές ότι είναι απαραίτητη μια καλή συνεργασία στην περιοχή αυτή και αυτό είναι προαπαιτούμενο για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στα θέματα αυτά. Έχουμε ζητήσει επίσης από τις τουρκικές αρχές να μην προβαίνουν σε προκλητικές δράσεις. Αυτά νομίζω τα, θα τα βρείτε και στις πρόσφατες απαντήσεις που έχω δώσει σε ώρα των ερωτήσεων. Συνεχίζουν οι συζητήσεις, υπάρχει εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πού βρίσκονται γιατί συνεχίζονται, αλλά ακολουθούν την, την φυσιολογική διαδικασία και για να απαντήσω στο ερώτημά μας έχουμε συζητήσει με την Σενεγάλη το πράσινο ακροτήριο και έχουμε προχωρήσει αλλά όχι με μεγάλη πρόοδο με το Μαρόκο, την Αίγυπτο και τη Μαυριτανία. Είναι οι φυσιολογικές λοιπόν διαδικασίες οι οποία γίνονται μέσω της Frontex. Το Συμβουλίο της Frontex παίρνει εντολή να ξεκινήσει αυτές τις συζητήσεις. Είχαμε επιτυχή συνεργασία με τη Ρωσία, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, αλλά λιγότερη πρόοδο με άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Προέρχεται από τον κύριο Κέλλη και αφορά τι διαπραγματεύσει για το κλίμα στην Κοπενχάγη. Υπουργό. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, που είστε, μάλιστα. Οι εξελίξεις ε, υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα προσπαθήσω να σα ενημερώσω για τις τελευταίες. Υπάρχουν δύο μείζωνα θέματα, ο μετριασμός και η χρηματοδότηση. Όπως είπε ο Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί, έχουμε ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε επιτυχή τελεσφόρηση στην Κοπενχάγη ε, που θα μας κρατήσει την αύξηση της θερμοκρασίας ε, κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου πριν από την, ε, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Εμείς παίζουμε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ούτως ώστε να φτάσουμε τελικά σε νομικά δεσμευτική συμφωνία. Τώρα θα έχουμε μια πολιτικά δεσμευτική συμφωνία σε μια πρώτη φάση και αργότερα θα περάσουμε ε, σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την περίοδο που ξεκινάει από την 1η Πρώτου 2013. Για να υπάρξει όμως συμφωνία θα πρέπει να έχουμε σύγκληση στα εξή θέματα. Καταρχάς, ε, βασικέ και φιλόδοξες ε, δεσμεύσεις μείωση από τι χώρε μέχρι το 2020. Η Ιαπωνία και η Νορβηγία έχουν κάνει κάποιες δεσμεύσεις, αλλά αυτό που υπάρχει επιτάπητος δεν είναι ικανοποιητικό για να πετύχουμε το στόχο των δύο βαθμών. Ε, γι' αυτό θα στραφούμε προς τις αναπτυγμένες συγγνώμη, χώρες, ώστε να έχουμε ε, και δράσεις και από τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, με, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Ινδονησία, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα συζητάνε αυτά τα θέματα. Αλλά η Κίνα και η Ινδία σίγουρα θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω δράσεις. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την αύξηση στους δύο βαθμούς. Γι' αυτό θα πρέπει οι προσπάθειες να γίνουν μεγαλύτερες, να αυξηθούν. Επίσης θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο για προσαρμογή στις ε, προσαρμογές, παραδείγματος χάρη μεταφορά τεχνολογίας και δυναμικού. Και χρηματοδότηση ε, με ένα σύστημα δίκαιο για το μετριασμό, την προσαρμογή οικοδόμηση δυναμικού και μεταφορά τεχνολογίας στι αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, ε, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, μιλήσαμε για τα τρία πρώτα χρόνια ότι θα έχουμε μια χρηματοδότηση για να υπάρξει μια ορμή στις διαπραγματεύσεις και να αυξηθεί η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων τώρα πλησιάζουν προς την Κοπενχάγη και ελπίζουμε ότι θα δώσουν ε, την πολιτική αυτή όφηση για τα βασικά θέματα του μετριασμού και τη χρηματοδότηση. Και θα υπάρξει, ελπίζω, μια φιλόδοξη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προ... υποβάλει προτάσεις για την περίοδο 2013 ε, ε, για να υπάρξει συμφωνία νομικά δεσμευτική. Τώρα, αν θα επιτευχθεί αυτό, είναι πολύ νωρί να το πω. Αλλά θα πρέπει να τα καταφέρουμε έξι μήνες ε, μετά την ολοκλήρωση τη διάσκεψης Κοπενχάγης. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μέλστρομ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συντομία και συνεκτικότητα της απάντησής σας, όχι μόνο στο δικό μου ερώτημα, αλλά σε όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο Κοινοβούλιο από τότε που εκπροσωπείται τη Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού των τη κίνα του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κοπεχάγη, κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο στο παρελθόν. Ποιο θα είναι ο τρόπο λειτουργία μια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή αν επιτευχθεί. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κύριε Κέλλη. <clears throat> σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Θα ξεκινήσουν αύριο οι πραγματικέ πολιτικές ε, διαπραγματεύσει με πρωθυπουργού και πρόεδρου από όλα τα κράτη τη Ευρώπη. Δεν πρέπει να μιλάμε για ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε να υπάρξει απαραίτητη δυναμική για μια γενική προσήλωση, για μια δεσμεύση όλων. Αν δεν επιτευχθεί, πρέπει να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσει. Δεν πρέπει εμεί να παρατήσουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ. Είναι το πιο σημαντικό θέμα στη γενιά μα. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Αν δεν υπάρχει συμφωνία αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο, θα πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι και να βρούμε μια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που έρχεται που έρχεται από τον κύριο Κέι Μίτσελ και αφορά την κλιματική αλλαγή και τη χρηματοδότηση για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το ίδιο θέμα είναι. Όπως είπε και ο βουλευτής, η χρηματοδότηση του κλίματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι τεράστιο θέμα για τις διαπραγματεύσεις στην Κοπενχάγη και θα είναι το κλειδί για να επιτευχθεί η οποιαδήποτε συμφωνία. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν πάρα αυτά δράσεις και να προετοιμάσουμε συλλογικές δράσεις ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και στο, στη Σύνοδο Κορυφή ε, του Δεκεμβρίου, πριν από λίγε μέρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είπαν ότι είναι έτοιμα για να δώσουν 2,4 εκατομμύρια ε, το χρόνο από τα χρόνια 2010 με 2012 για να βοηθήσουν αναπτυσσόμενες χώρες για να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος. Νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ένα, στενό, ένα ισχυρό μήνυμα στους διαπραγματευτές, διαπραγματευτές και αυξάμε την αξιοπιστία μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μέχρι το 2020. Θα πρέπει η σημερινή αρχιτεκτονική δομή να αναθεωρηθεί και να υπάρξουν μεταρρυθμίσει, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει. Όπω είπατε στο ερώτημά σα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου επικύρωσε τα όσα είπε η Κομισιόν, ε, γιατί είπε ότι το κόστο προσαρμογή θα μπορούσε να είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 2020. Ε, θα πρέπει οι αναπτυσσόμενε χώρε να κάνουν τι προσπάθειε του, να υπάρξει διεθνή δημόσια χρηματοδότηση. Και αυτό είναι μια εκτίμηση που κάνουμε. Δεν είναι προσφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλε εκτιμήσει από άλλε πηγέ. Αυτή είναι η εκτίμηση τη Κομισιόν. Ε, το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φω και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Συνολικά, θεωρούμε ε, ότι ε, κάθε χρόνο θα χρειάζονται 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 2020 δημόσια στήριξη τουλάχιστον. Και όλες ε, οι χώρες θα πρέπει να συνεισφέρουν μέσω σε αυτό το σύστημα ανάλογα με το ΑΕΠ τους και οι πιο φτωχές ακόμα χώρες. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει εμείς, οι αναπτυσμένες χώρες, ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο ώστε να μην επιτρέψουμε μια αύξηση πάνω από δύο βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ όπως και ο κύριος Κέλλη θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ποιότητα των απαντήσεων της κυρίας Υπουργού και γενικά για την ποιότητα της Σουηδικής Προεδρίας. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Υπουργό. Μας είπανε ότι θα είναι ο πρόεδρο των ΗΠΑ στην Κοπεχάκη και ότι είναι σε επίπεδο συζητήσεων με ηγέτες αναπτυσσομένων χωρών. Το έχει, έχει συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συζητήσεις και έχει προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα με τις ΗΠΑ και άλλους για να μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία στην Κοπεχάγη. Θα μπορούσε κύριε Υπουργό να διαβεβαιώσει το Κοινοβούλιο ότι αν υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση για τον αναπτυσσόμενο κόσμο θα είναι νέα χρήματα και όχι χρήματα τα οποία υπάρχουν ήδη στην αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της πείνας. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Πρώτο ερώτημα. Το φινόπορο έγιναν πολλές διμερείς επαφές για να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τις, και να προετοιμάσουμε τι διαπραγματεύσει. Είμαστε σε συνεχεί επαφές με τις ΗΠΑ για να σπρώξουμε και να περάσουμε ε, μία πιο φιλόδοξη δήλωση από αυτέ. Ε, σε ορισμένε από αυτέ τι διμερεί επαφέ, ε, εμπλακήκαμε πιο πολύ Είχαμε έξι διμερείς επαφές επί Σουηδικής ε, με την Κίνα, Ινδία, ε, Ουκρανία, Νότια Αφρική, Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν. Και οι κλιματικές αλλαγές ήταν πάνω, πάνω στην ατζέντα. Ε, είχαμε πολλές λοιπόν συνεδριάσεις για τη χρηματοδότηση. Είναι ένα συνδυασμός ε, παλιών και καινούριων χρημάτων. Κάποιες χώρες έχουν προτείνει ένα μείγμα, κάποιες άλλες ε, έχουν ε, κρατήσει ένα τμήμα τη αναπτυξιακής του βοήθειας για το κλίμα εδώ και κάποια χρόνια και επίση οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε είναι αυτέ που θα πληγούν περισσότερο από το, κλιματικέ κλιματικές αλλαγές. Και επομένω, το λογικό είναι ένα τμήμα του αναπτυξιακού προπολογισμού να πάει συγκεκριμένα για διάφορε κλιματικέ δράσει. Ω συνέπεια τώρα τη οικονομική κρίση, βέβαια, πολλά κράτη-μέλη δυστυχώ έχουν μειώσει τι φιλοδοξίε του στο συνολικό αναπτυξιακό προπολογισμό και αυτό είναι κρίμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα μείγμα πούμε, από δράση και από μέτρα και από χρηματοδότηση. Αλλά οφείλεται και στην κρίση. Και τώρα περνάμε στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Αντάμ Κόσα και αφορά την πρόταση οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεπιθήσεων αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Κύριε Υπουργέ. Eh, ευχαριστώ. Τα μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση είναι υψίστης σημασίας για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις. Όπως ε, λέει και ο αξιότιμος βουλευτής ε, στην ε, ερώτησή του. Επί Σουηδικής Προεδρίας προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι τεχνικές διατάξεις της οδηγίας για την ίση μεταχείριση. Υπάρχουν ή τέσσερις βάσεις διακρίσεων που δεν καλύπτει το κείμενο. Ε, θρησκεία, πεπιθήσεις, ε, ηλικία και σεξουαλικός προσανατολισμός. Στις 30 Νοεμβρίου υιοθετήσαμε μία έκθεση ως Προεδρία σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, το πεδίο τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων. Η Προεδρία επίσης αναφέρει ότι το ειδικό θέμα της παραγωγής αγαθών θα πρέπει να καλύπτεται από την πρόταση και θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Επίσης λέμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να επιληθούν σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις της οδηγίας. Και για να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία θα πρέπει να επιτύχουμε ένα κείμενο το οποίο να βρίσκει σύμφωνα όλα τα κρατημέλη. Ε, όλα τα κρατημέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσει και οι συζητήσει για την εφαρμογή και την ημερομηνία εφαρμογή καθώς και το πεδίο ε, δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ κύριο Σκόζα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την απάντησή της. Βλέπω ότι έχουν γίνει ορισμένα πρώτα βήματα τα οποία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν 50 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν αναπηρία. Αυτό το θέμα δεν αφορά μονάχα τους, τους ε, νέους. Είναι μια κοινωνία που γυράσκει με τρόπο ευτυχή η ευρωπαϊκή κοινωνία. Δεν είναι μονάχα τα άτομα λοιπόν τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν σε νεαρή ηλικία αναπηρίες, αλλά και τα άτομα τα οποία σε μεγαλύτερη ηλικία θα χρειαστούν αναπηρικά καροτσάκια και διευκολύνσεις για πρόσβαση στα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στις υπηρεσίες, η καταληκτική προθεσμία των 10 ετών αναφέρθηκε προηγουμένως και είναι πολύ σημαντικό να την τηρήσουμε γιατί είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Υπουργός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με το έντιμο μέλος για την ανάγκη να υπάρξει μια τέτοια οδηγία. Υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες της καθημερινής ζωής και έχουν επομένως προσκόμματα στην ελευθερία τους και την δυνατότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Λυπάμαι λοιπόν πολύ για αυτό το γεγονός. Το Συμβούλιο συζητά τα θέματα αυτά Χρειάζεται πολλή χρόνο βέβαια για τι συζητήσει αυτέ, γιατί είναι ρηξικέλευτη αυτή η πρόταση η οποία θα διατυπωθεί και έχει σημαντικέ κοινωνικέ και χρηματοοικονομικέ συνέπειε. Θα χρειαστεί λοιπόν η συνένεση όλων των κρατών μελών και στη συνέχεια, προτού εγκριθεί αυτή η οδηγία, θα πρέπει να περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάναμε διαπραγματεύσει σε μία σειρά ομάδων εργασία στο Συμβούλιο. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο Πρέπει όμω να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα το επίπεδο συνένεση που απαιτείται. Θα συνεχίσουμε όμω τι προσπάθειέ μα μέχρι το τέλο τη θητεία μα <clears throat> και πιστεύω ότι και η Ισπανική Προεδρία που θα πάρει τη σκητάλη θα, θα πράξει ό,τι μπορεί για να επιτύχει μια λύση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ. Περνάμε με το θέμα τη κυρία Πλινκεβίτσιουτε σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε τις κοινωνικές δυσκολίες που είναι και αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Φυσικά είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε ομάδες του πληθυσμού που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς και πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε και τον αποκλεισμό. Ξέρουμε ότι τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευπαθείς ομάδες δεν είναι σε θέση να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή λόγω των διακρίσεων. Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία του να τους εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην αγορά εργασίας από τους ανθρώπους. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας και έχουμε και κατευθυντήριες γραμμές. Ε, το Μάρτιο του 2008 ε, το Συμβούλιο ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία Τη ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία, αναφέρεται ε, στα συμπεράσματα τη 20 Νοεμβρίου 2009 του Συμβουλίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασία. Είναι προϋπόθεση και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή μας. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκαναν μια κοινή συμφωνία ότι το 2010 θα είναι η χρονιά για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να συμπεριλάβει και την έννοια του εκπαίδευση για όλους και ίση πρόσβαση στην τεχνολογία. Για όλους και κυρίως για άτομα με αναπηρίες. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία και άλλους μειονεκτούντες ανθρώπους. Επίση, περιμένουμε και άλλε πρωτοβουλίε να προωθηθούν ε, μέσα στο ίδιο πνεύμα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση των ε, ατόμων ανεξάρτητα από τη θρησκεία πεποίθηση, την ηλικία ή του ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες θα επηρεαστούν θετικά αν γίνει πραγματικότητα η του σεξουαλικου προσανατολισμου πιστευουμε οτι οι ανθρωποι με αναπηριε θα επηρεαστουν θετικα αν γινει πραγματικοτητα η προταση της Κομισιόν. Και η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τις κοινωνικές υποθέσεις ασχολείται ακόμα με το κείμενο αυτό στις διάφορες συζητήσεις της. Υπάρχει και μια έκθεση προόδου που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο, αλλά δυστυχώ δεν έχει επιτευχθεί ακόμα κοινή συμφωνία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα ακόμα από αυτέ τι διαπραγματεύσει, οι οποίες είναι εν εξελίξη. Θέλουμε να προκύψει ένα καλό κείμενο φυσικά. Και όπως ανέφερα, τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν για αυτή την πρόταση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δουν ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη οικονομική κρίση σε αυτό το πλαίσιο και για αυτού του ανθρώπου. Αλλά άπαξ και υπάρξει ομοφωνία, φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα το ενθαρρύνουμε ε, με βάση τη συνθήκη τη ε, Λισαβόνα να υποστηρίξει και αυτό το μέτρο που θα προκύψει. Η κυρία Πλυνκεβισιούτε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Υπουργό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σουηδία εν γέννη, γιατί επί Σουηδικής Προεδρίας το Συμβούλιο Υπουργών ε, προσυπέγραψε την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό είναι μια καλό, ένα καλό βήμα, αλλά απλώς ένα βήμα. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές πραγματικότητες. Σε ορισμένα Ορισμένοι ανάπηροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν καν τη νοηματική γλώσσα. Ε, σε άλλα κρατημέλη υπάρχουν άλλες ελλείψεις. Μην ξεχνάμε ότι περίπου το 10% των πολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάπηροι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, στην εφαρμογή της οδηγίας κατά των διακρίσεων, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να προωθήσουμε μια χωριστή οδηγία για τα δικαιώματα των αναπήρων, που θα είναι δεσμευτική για όλους μας και που θα εμποδίζει την πρόθεση των διακρίσεων των ατόμων με αναπηρία. Υπουργό. Νόμιζα ότι υπήρχε και άλλο ερώτημα. Ας υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για έλλειψη πολιτικής θέλησης. Κατανοούμε την σημασία αυτής της οδηγίας και έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Δεν μπορώ να αλλάξω το γεγονός ότι απαιτείται ακόμα ομοφωνία στο Συμβούλιο και η, η ομοφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Η Σουηδική Προεδρία έχει προσπαθήσει να προτείνει διάφορες ε, συμβαστικές λύσεις. Υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας οι οποίες εργάζονται και εξακολουθούν αυτές οι συνεδριάσεις αυτών των ομάδων εργασίας ενώ συζητούμε σήμερα μέχρι το τέλος της Προεδρίας θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν δεν επιτύχαμε ακόμα μια ομοφωνία κρίμα θα είναι να κόψουμε σε κομμάτι αυτή την οδηγία γιατί ο στόχος μας και αυτό, σε αυτό μας ενθάρρυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να έχουμε μια συνολική οδηγία για τις διακρίσεις αν αρχίσουμε να αποσπούμε κομμάτια δεξιά και κομμάτια αριστερά, θα χαθεί αυτή η συνολική ε, αντιμετώπιση τη οδηγία. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να επιτύχουμε μια έγκριση όλη τη οδηγία, γιατί αυτό θα είναι κεφαλαιόδε για τον αγώνα κατά των διακρίσεων κατά των αναπήρων, αλλά κατά όλων των θυμάτων διάκριση. Ευχαριστώ, κυρία. Ε, Πρόεδρε, οι συμπληρωματικέ ερωτήσει έχουν χρόνο 30 δευτερόλεπτα, όχι ένα λεπτό. Έχω κάποιε αιτήσει συμπληρωματικών ερωτήσεων για αυτό το ερώτημα. Πρέπει να λάβω υπόψη το γεγονό ότι υπήρξε μια σειρά με την οποία ζήτησαν το λόγο διάφοροι συνάδελφοι και το αν μίλησαν ή δεν μίλησαν στο παρελθόν. Η κυρία Κλάς και η κυρία Μακίνες, θα λάβουν το λόγο. Λοιπόν, η κυρία Κλάς πρώτη. Χωρίς μικρόφωνο. Κυρία Πρόεδρε, προφανές θα πρέπει, είναι ότι πρέπει να εμποδίσουμε τις ε, διακρίσεις. Όλοι μας πρέπει να το πράξουμε αυτό. Συμφωνείτε μαζί μου κυρία Πρόεδρε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σαφείς γνώμονες για το πώς μπορεί κανείς να ορίσει μία διάκριση. Παραδείγματο χάρη, κάποιο νοικιάζει ένα σπίτι και δεν θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι και δεν τα καταφέρνει και καταγγέλει ότι υπήρξε διάκριση εναντίον του. Μήπω θα πρέπει η Κομισιόν. <clears throat> Μήπως θα πρέπει να υπάρξει μια αίτηση προ τα κράτη-μέλη να διευκρινίσουν τι εθνικέ του διατάξει, Γιατί είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν κοινέ ρυθμίσει στα θέματα διακρίσεων σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Μαχ εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου. Εφόσον μιλάμε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο κύριος Κότσα εξελέγει πρόσφατα πρόεδρος της διαπαραταξιακής ομάδας για τους αναπήρους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την οικονομική κρίση. Είχαμε μια συζήτηση χθε και νεύεται καταφατικός μας ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα της ε, ε φροντίδας των παιδιών σε, θεσμι... ιδρύματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τύχει μεγάλη προσοχή και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να κινδυνεύσει από την οικονομική κρίση. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καιρού κρίσεων πάντα φύγονται οι πιο τροτοί. Νέοι, γέροι, άνθρωποι με, ειδικά, ε, με, και επομένως θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και έχει προσταθεί στα συμπεράσματα διαφόρων συμβουλίων, καθώ και στι συστάσεις που προκύπτουν και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη το γεγονό ότι πιο ευπαθεί ομάδε είναι εκείνε που πλήττονται περισσότερο και βασανίζονται περισσότερο. Συμφωνώ λοιπόν, προφανώ με αυτό. Και ω απάντηση στο ερώτημά σα, θέλω να σα πω ότι πριν προκύψει η σφαιρική οδηγία, ε, δεν μπορούμε να θέσουμε πρότυπα ευρωπαϊκού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις προς τους ανθρώπου ανθρώπους με αναπηρία. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική σφαιρική οδηγία και μετά με βάση αυτή να δουλέψουμε. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει τεράστια προσπάθεια, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν μαζικές διακρίσεις, ε, μαζικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή του ζωή οι ανάπηροι και τους εμποδίζει να ζήσουν φυσιολογικά και να εκπληρώσουν το δυναμικό τους. Νομίζω όμως ότι πρέπει πρώτα να φτιάξουμε μια οδηγία και συνεχεία να δουλέψουμε και να υποφεληθούμε από την ε, επόμενη χρονιά, που είναι η χρονιά κατά πολέμηση του αποκλεισμού ε, και να οργανώσουμε διάφορε κοινέ εκδηλώσει, ούτω ώστε να υπάρξει αφύπνιση σε όλα τα κρατημέλη για αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ε, είμαι πεπισμένη ότι στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να συγχαρώ και τον κύριο Καζάν για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου τη διαπαραταξιακή. Πάμε πολύ γρήγορα στις επόμενες ερωτήσεις. Οι 8 και οι 9 έχουν ε, αποσυρθεί. Οι 10 δεν είναι παραδεκτή, γιατί ήταν αντικείμενο χωριστή συζήτηση ε, που κάναμε σήμερα. Επομένως, τώρα πάμε στην ερώτηση 11 του κ. Παλέκης, που δεν είναι όμως παρόν και επομένως δεν συζητείται. Και επομένως πάμε στο ερώτημα του κ. Αγκουράκη για τις φρικαλές δολοφονίες φτωχών περουβιανών αγροτών με σκοπό το κέρδος. Κύριε Υπουργέ, αν είσαστε έτοιμοι, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μία από τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωση, από τις αξίες που προωθούμε. Και το Συμβούλιο βεβαίω γνωρίζει ότι σε όλε τι σχέσει μα με τι τρίτε χώρε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο γεγονό που αναφέρει ο βουλευτή, στο Συμβούλιο δεν το συζητήσαμε, δεν το ξέραμε. Φυσικά είχαμε διαβάσει τα δημοσιεύματα του τύπου, αλλά σημειώνουμε ότι οι πιο πρόσφατες ε, εκθέσεις λένε ότι ίσως η αρχική ιστορία, τα αρχικά δημοσιεύματα, ίσως δεν ήταν ακριβή. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε απλά δημοσιεύματα του τύπου ως Συμβούλιο. Επομένως, η Σουηδική Προεδρία δεν μπορεί να αντιδράσει ούτε καν να εκατολογήσει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Σαγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι δεν με ικανοποιεί καθόλου η απάντηση ε, της ε, κυρίας Υπουργού πρόκειται για ένα φρικαλαίο έγκλημα για ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο θα έλεγα και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή ένωση όταν θέλει έχει εκείνα τα μέσα ώστε να διερευνήσει ε, πιο εμπεριστατωμένα τα ζητήματα αυτά τέτοιας φύσης και επειδή υπάρχουν και οι σχέσεις με το περού απαιτούμε να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση εκ μέρους ε, της κυβέρνησης του περού για το συγκεκριμένο περιστατικό και να υπάρχουν μέτρα αλλιώς θα βλέπουν να επαναλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις. ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε αντικρουόμενες εκθέσεις για το θέμα αυτό από διάφορες αρχές και σε ό,τι αφορά τα δημοσίευματα στον τύπο. Φαίνεται ότι δεν είναι βάσιμες αυτές οι οι αναφορές για αυτά τα γεγονότα. Εάν είχαν λάβει χώρα αυτά τα γεγονότα θα ήταν πράγματι φρικτά. Αλλά μπορεί αυτά τα δημοσιεύματα να είναι μη ακριβή και εμείς ούτως ή άλλως δεν έχουμε την αρμοδιότητα να αντιδράσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ερχόμαστε στο ερώτημα του κυρίου Τσαρνέσκι και αφορά τη διάκριση τη διακρίση σε βάρος της πολωνικής μειονότητας στη Λιθουανία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δίνει μεγάλη προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναφέρεται εξάλλου και στη Χάρτα των Θεμελιωδών και στην Ιδρυτική Συνθήκη και θα συνεχίσει να επιμένει στην παρακολούθηση και καταδίκη όλων των τύπων διακριτικής μεταχείρισης. Το θέμα της προστασίας των μειονοτήτων επίσης ε, το συζητάει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τις εθνικές μειονότητες. Το θέμα που έθεσε η κυρία Χανέκε εξετάζεται αυτή τη στιγμή μάλιστα από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον Ιούνιο του 2000 έχει εγκριθεί, είχε εγκριθεί η οδηγία για την ίση μεταχείριση που απαγορεύει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση με βάση θρησκεία κλπ και συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένους τομείς ε, εργασίας προστασία σε κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Και καθήκον της Κομισιόν είναι να παρακολουθεί κατά πόσον εφαρμόζονται όλα αυτά σωστά. Τέλος, στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου φέτος, η ανάγκη για πρόσθετες προτάσεις για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες έχει συζητηθεί με βάση τη συνθήκη της Χάγης η συντάσουσα ή η συντάξασα ο συντάξας μάλλον ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την απάντησή σας και ιδιαίτερα γιατί τονίσατε ότι το Συμβούλιο καταδικάζει κάθε μορφή άνησης μεταχείρισης ή διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των οποίων και των εθνικών μειονοτήτων όπως την πολωνική μειονότητα στη Λιθουανία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ελπίζω και οι λιθουανικές αρχές να συμμορφωθούν γιατί παραβιάζουν συνεχώς τα δικαιώματα της μειονότητας σε θέματα παιδείας και αλέως. Παρακαλώ λοιπόν να παρακολουθείτε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τις αρχές και αξίες που αντιπροσωπεύει η Ένωση και άρα και το Συμβούλιο και τα συγκεκριμένα γεγονότα που ανέφερε η ερώτηση. Εξετάζονται, είπα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν σημειωθούν κι άλλες μορφές διακριτικής ή άνησης μεταχείρισης, θα φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τις συνθήκες και με τα στην Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Ο κύριος Γκάλαγκερ έφτασε, είδαμε χαρά μου, για να αντικαταστήσει τον κύριο Κρόλη για το επόμενο ερώτημα που αφορά την δίωξη ε, μοναχών στο Βιετνάμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα το Συμβούλιο γνωρίζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και των βουδιστών αυτών μοναχών την περίπτωση. Δύο φορές το χρόνο η Κομισιόν και το Συμβούλιο κάνουν μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις χώρες αυτές. Η τελευταία έγινε στις 11 Δεκεμβρίου στο Ανόη και συζητήθηκαν θέματα ελεύθερης έκφρασης, και των δικών που γίνονται εκεί ως προς την ελευθερία της άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Για συγκεκριμένους ε, κρατουμένους συζητήθηκαν επίσης περιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε τα ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα με τους βουδιστές μοναχούς. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν επίσης συζήτησαν διαμα με τους ε, κατοίκους ενός χωριού και ανέφεραν τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο. Έγιναν συναντήσεις εκπροσώπων της Κομισιόν με υψηλού επίπεδου αξιωματούχους του κυβέρνηση του Βιετνάμ και οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν του χρόνου. Εκφράσαμε πάντως σαφώς ε, τις απόψεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ την προ... συζητήσαμε για προστασία της περιουσίας εκκλησιών. Αυτά τα ξέρει το Κοινοβούλιο, αλλά μιλήσαμε και ιδιαίτερα για την κατάσταση στο χωριό εκείνο πλάν. Και τονίσαμε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των μονομένων συμβάσεων που έχει συνυπογράψει το Βιετνάμ. Σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ, μάλλον χάρη στο ψήφισμα αυτό, έχουμε κατευθυντήριε γραμμές να ακολουθούμε και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να παίξει ισχυρότερο ρόλο στο μέλλον για την κατάσταση στο Βιετνάμ 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε μοναστήρια πάλι στο χωριό αυτό το Πλάνναμ και είδαμε τι συμβαίνει εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, την κυρία Υπουργό για την πλήρη απάντησή της. Και θα ήθελα όμως, του κύριου Κρόουλε να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την προσέγγιση και του Συμβουλίου και τη Κομισιόν και θα συνεχίσουμε με πραγματιστικό τρόπο να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη πρόταση, άλλη αίτηση για λήψη του λόγου. Περνάμε στο επόμενο ερώτημα που είναι αυτή τη φορά από τον κύριο Γκάλαχερ και αφορά την αίτηση της Ισλανδίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό είναι ένα ερώτημα και για σας πιστεύω. Έντιμε κύριε Γκάλαχερ, θα σας υπενθυμίσω ότι είπανε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 10 και 11 Δεκεμβρίου. Είπαν ότι η Ισλανδία είναι μια χώρα με παλιές και βαθιές δημοκρατικές δομές και αξίες. Έχει μεγάλη δυνατότητα να συμβάλλει τα μάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικά και στρατηγικά. Είναι πολύ στενά ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομεί λόγω τη παρουσίας τη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική ε, Περιοχή και στη ζώνη του Σέγγεν. Η αίτηση της, ε, ε της Ισλανδίας υπευλήθη στην Σουηδική Προεδρία στις 16 Ιουλίου 2001. Στην υποφαινόμενη μάλιστα υπευλήθη αυτή η αίτηση. Στις 27 Ιουλίου στη συνεδρίασή του το Συμβούλιο συμπεφώνησε ότι μπορεί να λάβει χώρα αυτή η η προσχώρηση βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου το 2006 που λέει ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει των ιδιαίτερων στοιχείων τους. Αποφασίσαμε ότι βάσει του άρθρου 49 της Συνδίκης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διεκπαιρεώσουμε την αίτηση της Ισλανδίας. Τώρα η Κομισιόν θα πρέπει να μας δώσει μια γνωμοδότηση σε σχέση με αυτή την αίτηση η οποία θα αντιμετωπιστεί βάσει των συνδικών και αυτό είχε ήδη αποφασιστεί στην Κοπεχάη του 1993 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2006. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων λοιπόν του Συμβουλίου, το θέμα αυτό θα συζητηθεί και πάλι από, από τη στιγμή που η Κομισιόν θα έχει υποβάλει την, αίτηση, την ε, γνωμοδότησή και το Συμβούλιο λοιπόν θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ισλανδία στους πρώτους μήνες της Ισπανικής Προεδρίας. Ο κύριος Γκάλαχερ. Μικρόφωνο κύριε Γκάλαχερ. Θα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Συμβουλίου για την απάντησή της και ως Πρόεδρος της αντιπροσωπείας η οποία αντιμετωπίζει το θέμα της Ισλανδίας κατανοώ πλήρω ότι βέβαια κάθε αίτηση πρέπει να αντιμετωπιστεί επί τη βάση των δικών της στοιχείων και της πρόοδου η οποία θα έχει επιτελεστεί αλλά είναι γεγονός ότι η Ισλανδία απήντησε σε πολλά ερωτήματα μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο ήταν πολύ θετικό, το ότι ήταν βέβαια και μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αυτό δείχνει την προσήλωση της Ισλανδίας για την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσουν τα σύνορά μας μέχρι την ακριτική Ισλανδία. Αλλά εν καιρό και εν κατακλείδη είναι μία από τις παλαιότερες δημοκρατίες της Ευρώπης και πρέπει οι πολίτες αυτής της δημοκρατίας να πάρουν την αντίστοιχη απόφαση. Εγώ προσβλέπω σε περαιτέρω πρόοδο στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου και ελπίζω ότι θα υπάρξει και ένα νέο θετικό βήμα και θα υπάρξει η αντίστοιχη ανακοίνωση από το Συμβουλίο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όλες οι διαδικασίες θα εφαρμοστούν. Πρέπει να διεκπαιρεωθεί έτσι η αίτηση της Ισλανδίας. Δεν έχει τελειώσει η εκπόνηση της γνωμοδότησης από την Κομισιόν μετά από τη διαδικασία του screening. Έχουν όμως ξεκινήσει οι Ισλανδοί να δημιουργούν ομάδες διαπραγμάτευσης και είναι έτοιμοι να κάνουν μια ταχεία διαπραγμάτευση για τα θέματα αυτά και οι δύο πλευρές. Μπορούμε να περιμένουμε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της στην αρχή του επερχόμενου έτους και ελπίσουμε ότι το Συμβουλίο μπορεί να πάρει τις αποφάσεις για περαιτέρω μέτρα το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Θα έπρεπε τώρα να εξετάσουμε το, το ερώτημα του κυρίου Ντερόσα, ο οποίος δεν είναι παρόν. Παίρναμε στο ερώτημα του, της κυρίας Μαχγκίνες για τα βιοδιασπόμενα απόβλητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε μέρα παράγουμε τεράστια ποσά αποβλήτων στα κράτη-μέλη. Πώ θα αντιμετωπίσουμε. Ο τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε έχει τεράστιε επιπτώσει στο περιβάλλον προφανώ. Στην πρόσφατη έκθεση τη Κομισιόν για την εφαρμογή τη ε, κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, βλέπουμε ότι διάφορα κράτη-μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολλά άλλα κράτη-μέλη για να υπάρξει κατάλληλη υποδομή για τη διαχείριση των αποβλήτων με βάση την οδηγία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις χωματερές. Το θέμα των υγειονομικών ταφών πρέπει να το δούμε. Ε, εννέα χώρες ε, έχουν εφαρμόσει τους στόχους του 2006. Τον Ιούνιο του 2009 τα συμπράσματα του Συμβουλίου ε, δήλωσαν ότι συμφωνούμε ο Συμβούλιο με την Κομισιόν και είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι ε, να υλοποιηθούν για τα βιοδιασπόμενα απόβλητα. Θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε μια αξιολόγηση ε, της νομοθεσίας για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα επίπεδα των αποβλήτων, όσο, όπου γίνεται βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση των βιοδιασπόμενων αποβλήτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα απόβλητα για τις εγκαταστάσεις ε, βιοαερίου, το Συμβούλιο επίσης ε, λέει ότι η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων θα μας οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των ε, αποβλήτων, ε, θα βοηθήσουμε έτσι το περιβάλλον και θα υλοποιήσουμε τους στόχους για την, το να μην χρησιμοποιούμε, να μην καταλήγουν τα βιοδιασπόμενα απόβλητα στις χωματερές. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Φυσικά σας υποστηρίζουμε, αν έχετε ποτέ σταθεί ε, στο χείλο μια χωματερή και έχετε εισπνεύσει, είναι φρικόδηση ως Ε, νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν τι σημαίνει χωματερή και όσα δεν τι έχουν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί μόνο εννέα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής έχουν ε, σεβαστεί τους στόχους. Πρέπει να προχωρήσουμε. Και ξέρω ότι πρέπει να προχωρήσουμε το βιοαέριο. Ε, όλοι συμφωνούμε με τις αρχές, αλλά γιατί δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε τους στόχους. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονε για αυτό το θέμα, αλλά αν κατάλαβα καλά από τη δήλωση τη Κομισιόν, δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή ε, σε κάποια κρατημέλη. Κοστίζει και πολύ να δημιουργηθεί. Φυσικά, μακροπρόθεσμα είναι υποφελέ. Αλλά τα κράτη-μέλη συχνά δεν επενδύουν για να υπάρξει κατάλληλη υποδομή, γι' αυτό ακριβώ καθυστερούμε τόσο πολύ. Τώρα θα πάμε στη τελευταία ερώτηση για σήμερα. Τώρα το τελευταίο ερώτημα, το τελευταίο ερώτημα της Προεδρίας σας από τον κύριο Hans Peter Μάρτεν. Επιτυχίες της Σουηδικής Προεδρίας του Συμβουλίου σε θέματα διαφάνειας. Νομίζω ότι εδώ έχετε να πείτε πολλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Σουηδία ως κράτος μέλος και για τη Σουηδία που έχει την ε, Προεδρία. Θα πρέπει να υπάρξει ε, ευρύτερη διαφάνεια, ε, μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα ήθελα να σας πω ότι η ιστοσελίδα της Προεδρίας του Συμβουλίου δίνει πληροφορίες για κείμενα, υπάρχει web streaming σε τρεις γλώσσες μάλιστα. Τους τελευταίους μήνες η Σουηδική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε για να βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα. Το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο είχαμε 20 δημόσιες συζητήσεις με την πρωτοβουλία ή υπό την αιγίδα της Σουηδικής Προεδρίας με βάση το άρθρο 8.3 του κανονισμού. Υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασία για το πρόγραμμα ECOFIN. Είχαμε 25 δημόσιε συζητήσει του τελευταίου μήνε στα πλαίσια του ECOFIN σε ό,τι αφορά τι ε, γενικέ ε, συζητήσει 59 ε, σημεία ε, έχουν συζητηθεί ως σημεία α και 9 ως σημεία β στη συζητήση του Συμβουλίου. Αν θεωρείτε ότι αυτά δεν είναι αρκετά, να μην ξεχνάτε τα σημεία στις συζητήσεις του Συμβουλίου που φτάνουν στο κοινό και που συζητούνται στα πλαίσια της συναπόφασης. Η νέα Επιτροπή σίγουρα θα αυξήσει τον αριθμό των νομοθετικών προτάσεων που θα συζητούνται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, όλες οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου για αυτά τα σημεία, τα νομοθετικά σημεία, θα είναι δημόσιες συζητήσεις. Και χαιρόμαστε βεβαίως για, για αυτό το γεγονός. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πιο δημοκρατική και πιο αποτελεσματική εξαιτία αυτού. Η... Χθες η Σουηδική Προεδρία υιοθέτησε μια πρωτοβουλία για να συναντηθούμε με τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για τη Διαφάνεια και η Μάρκοτ Βάλστρομ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η κυρία Γουόλιτς, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, συζήτησαν διάφορες πρακτικές προτάσεις για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην πληροφορία, στις πληροφορίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και να καταστήσουν αυτές τις πληροφορίες πιο φιλικές για τους ακροατές και για το κοινό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι συγκινητικό, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά το γεγονός ότι μπορώ να ανταλλάξω το τελευταίο ερώτημα της Προεδρίας σας μαζί σας κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Γνωρίζετε ότι πολλές φορές είναι τα μικρά βήματα τα οποία πολλές φορές πηγαίνουν σαλιγκαροδός από πλευρά ταχύτητος που μας έχουν οδηγήσει στην διαφάνεια η οποία υπάρχει σήμερα. Βέβαια οι ένθερμοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι με όλα αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί. Εμείς παραμένουμε με το μήνυμά σας ότι μπορεί ακόμα περισσότερο να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Εγώ σκέφτομαι τις ομάδες εργασίας των ειδικών ομάδων του Συμβουλίου όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια σε σχέση με την μέση διάταξη των εργασιών τους αλλά βλέπετε με μακροπρόθεσμη προοπτική να μπορέσουμε να φτάσουμε ως Ευρώπη εκεί που βρίσκεται ήδη η Σουηδία σε 10 χρόνια κυρία Υπουργό. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πρόσβαση στα έγγραφα και η διαφάνεια έχει βελτιωθεί πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό οφείλεται στον κανονισμό 1049 που είναι πάρα πολύ σημαντικός κανονισμός και χαίρομαι που συνέβαλα στην έγκριση αυτού του κανονισμού και επίσης είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό είναι πολλά άτομα τα οποία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχουν κατανοήσει ότι η διαφάνεια δεν είναι αρνητική αλλά θετική. Είναι πολύ καλή για την νομιμοποίηση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνει τις δυνατότητες να υπάρξει διαφθορά και ατασταλίες. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Μας δίνει νέες δυνατότητες στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζω ότι όλες οι επερχόμενες κατά σειρά προεδρία θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο στο μέλλον και υπεχθέσει η Κομισιόν ότι θα επανέλθει με προτάσεις οι οποίες θα εκκινούν από τη συνθήκη της Λισαβόνας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον στα θέματα της διαφάνειας. Πολλά παραμένουν να πράξουμε, αλλά έχουμε φτάσει ήδη ένα σημαντικό επίπεδο και όπως είπε το αξιότιμο μέλος είναι ένας συνεχής αγώνας και θέλω να το συνεχίσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο ερώτημα θα απαντηθεί εν τα άλλα ερωτήματα εκτός από το 19 που θεωρήθηκε απαράδεκτο θα απαντηθούν εγγράφως. Θέλω ευχαριστήσω την Υπουργό, αγαπητή Σεσίλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συχνή σου συμμετοχή στις συζητήσεις μας κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας και για τις απαντήσεις σου προσβλέπουμε να υπάρξει ε, και συνέχισα τη συνεργασία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ και σε εσά και την ομάδα σας. Έχει κλείσει λοιπόν η ώρα των ερωτήσεων. Η επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αύριο 5η 17 Δεκεμβρίου 2009 από τις 9 μέχρι, μέχρι τη 1 και από τις 3 μέχρι τη 5 έχει δημοσιευθεί η μέση διάταξη στο διαδίκτυο τέρμα συνεδρίασης.